του κυκλοφορία Σέγγεν. Να δώσουμε χέγγια στου πολίτε μα ότι μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε, λέει ο πρόεδρο. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά σα. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, που είναι και το τελευταίο απόψε και που είναι η προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με θέματα αθλητισμού. Ιδιαίτερα όσον αφορά του εκπροσώπου ποδοσφαιριστών, μάνατζερ ποδοσφαιριστών στην ημερήσια διάταξη εκπροσώπους ποδοσφαιριστών. Για την προφορική ερώτηση <clears throat> η κυρία Ντόρις Πάκα έχει τρία λεπτά για να παρουσιάσει αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Η κυρία Πάκα, πρόεδρε, αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη στην έκθεση η Βομπέλετ είχε αναφερθεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στην ανάγκη καλύτερης ρύθμισης ε, των ε, δραστηριοτήτων των μεσολαβητών ε, παικτών και των εκπροσώπων ποδοσφαιριστών. Και έχουμε τώρα αυτό το θέμα εδώ. Η νομική κατάσταση είναι συγκεχημένη. Πολλές φορές διασυνοριακά δραστηριοποιούνται αυτοί οι παίκτες και έτσι η εθνική νομοθεσία δεν είναι η πιο ενδεδειγμένη να ρυθμίζει αυτές τις δράσεις οι αθλητικές ενώσεις και οι λέσχες είναι περιορισμένες όσον αφορά τη δράση τους. Ως μη κρατική, ε, οι εκπρόσωποι δεν έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν αυτά τα θέματα αφ' αυτών. Η FIFA για παράδειγμα την ε, ε, διαδικασία και τις ρυθμίσεις για τους εκπροσώπους παικτών τις αποδυνάμωσε. Δημοσιεύθηκε μία μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα όσον αφορά ανησυχητικές ε, διασυνδέσεις εκπροσώπων επαγγελματιών παικτών και εγκληματιών. Μπορεί κανείς να κάνει λόγο εδώ για πλήσιμο χρήματος, φοροαπάτη, φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής. Τέτοιου είδους όμως ε, κατηγορίες ε, υπονομεύουν τα αθλήματα αυτά και δεν ευθυγραμμίζονται με τα κοινωνικά αιτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μελέτη της διαπιστώνουν ότι οι χρηματοοικονομικές ροές μεταφορών παικτών, εξαγορών παικτών είναι σε γίνονται σε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας και έτσι θα πρέπει εδώ να δούμε πάλι τα θέματα εγκληματικών συνεργών. Ιδιαίτερο όμως για την εκπροσώπηση νέων παικτών υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος. Εδώ νέοι άπειροι παίκτες αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ώστε για παράδειγμα από την Αφρική να τους δίνουν υποσχέσεις για μια μεγάλη σταδιοδρομία στην Ευρώπη και αν δεν βρίσκεται κάποια λέσχη να απασχοληθούν, τους εγκαταλείπουν και έτσι ως παράνομοι ε, μετανάστες αντιμετωπίζονται στην Ευρώπη. Εν ώψη αυτή τη κατάσταση, μια ευρωπαϊκή νομοθετική ρύθμιση απαιτείται. Έτσι, μια ενιαία ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργηθεί, θα κλείσουν τα παραθυράκια για την ε, υπονόμευση του νόμου και έτσι θα μπορέσει η ε, δραστηριοποίηση των εκπροσώπων παικτών να γίνεται σε ένα διαφανές πλαίσιο. Έτσι πρέπει να έχουμε ένα στόχο ώστε η μεταφορά ανήλικων παικτών να αποκλεί οποιαδήποτε πληρωμή ποσοστών μέσω διαμεσολαβητών, ώστε να μην υπάρχει κίνητρο για τέτοιου είδους αθέμητες πρακτικές όσον αφορά ανήλικους ε, ε, παίκτες. Ελπίζω ότι η πρότασή μας θα βρει την συνένεση στην Ολομέλεια και κυρίως θα δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ Ντόρις. Πάντα υπόδειγμα είσαστε στην χρήση του χρόνου. Πάντα είσαστε υποδειγματικοί. Θα λάβει τον λόγο η Επίτροπο, τώρα, Βασιλείου, η κυρία Βασιλείου, για να τοποθετηθεί εξ ονόματο τη Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πακ που υπέβαλε αυτή την προφορική ερώτηση εκ μέρου τη Επιτροπή Πολιτισμού. Ξέρω πολύ καλά την πολιτική σπουδαιότητα που έχει αυτό το θέμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μια ανεξάρτητη μελέτη για του μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση των όλων, ε, του όλου θέματος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου 6.000 μάναζερ που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη σε διάφορους τομείς. Όμως, 95% εξ αυτών δραστηριοποιούνται μόνο σε τέσσερα αθλήματα. Στο στίβο, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο ράγπι. Και στα πλαίσια αυτής της ομάδας το ποδόσφαιρο κυριαρχεί βεβαίω, σαφώ. Η μελέτη επίση αυτή μα λέει ότι μόνο ένα περιορισμένο αριθμό των κρατών μελών ε, έχουν κανονιστικέ ρυθμίσει για του μάνατζερ. Στι περισσότερε χώρε βασίζονται περισσότερο σε γενικού ε, κανόνε και διατάξει είτε του εργατικού δικαίου είτε του δικαίου γενικώ. Όμω, ε, πολλέ αθλητικέ ομοσπονδίε έχουν υιοθετήσει κανονισμού ε, για του μάνατζερ, όχι μόνο σε αυτού του τέσσερι τομεί που ανέφερα. Παρόλο που οι υπάρχοντες ε, δημόσιοι και ιδιωτικοί κανονισμοί μπορούν να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και να δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου, υπάρχουν ε, σύμφωνα με τη μελέτη ε, κάποια εμπόδια ε, για την ρύθμιση του θέματος αυτού. Η μελέτη επισημαίνει ε, αμφίβολης νομιμότητας ε, πρακτικές, παραδείγματος χάρη ε, μυστικές μίζες που καταβάλλονται, ε, εκμετάλλευση νέων αθλητών κλπ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά για να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα και την δικαιοσύνη των αθλητικών αγώνων ο αθλητικός κόσμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Γι' αυτό διάφορα ε, όργανα έχουν υιοθετήσει μέτρα για την ε, ρύθμιση των δραστηριοτήτων των μάνατζερ. Οι κανόνες αυτοί που μπορεί να έχουν κάποια πλέον πλεονεκτήματα. Οι αθλητικές κυρώσεις μερικές φορές είναι ε, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν αθέμικες ε, πρακτικές στην αγορά. Είτε από ομάδες, είτε από αθλητές, είτε από τους μάνατζερ. Όμως η αθλητική τα αθλητικά αυτά όργανα δεν έχουν την εξουσία να ε, κάνουν έρευνες και να τιμωρούν ε, πρακτικές όπως είναι η διαφθορά, η δωροδοκία, ε, η, το ξέπλυμα χρήματος και η παράνομη μετανάστευση. Το αθλητικό κίνημα λοιπόν ζητάει τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και εδώ η Κομισιόν έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Μπορούμε να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη κοινών αρχών και προτύπων που θα λειτουργήσουν σε ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων για όλε τι αθλητικέ ομοσπονδίε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τι είδου δράσει θα ήταν οι πιο σωστοί και κατάλληλοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διάφορε εναλλακτικέ ε, λύσει ε, κατά νου, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ποια δράση θα αναλάβουμε και για να γίνει αυτό χρειάζονται περαιτέρω διαβουλεύσεις ε, και συζητήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα παρέμβουν τώρα εξ ονόματο των ομάδων ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα για 3,5 λεπτά ο κύριο Μπέλετ, εξ ονόματο του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Απευθύνομαι στην κυρία Επίτροπο και ευχαριστώ που στείλατε ε, την, ε, που ασχοληθήκατε ε, με το κύπελο στην Νότια Αφρική. Βλέπουμε πόσο το ποδόσφαιρο είναι καλό για μια χώρα και για τη ζωή. Γενικά θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τον αθλητισμό από όλε τις εγκληματικέ συμπεριφορέ για τις οποίες μίλησε η κυρία Πακ και να καταβάλουμε προσπάθειες για να εξαλείψουμε τα προβλήματα. Στην μελέτη που αναφερθήκατε και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, διαβάζουμε ότι ο αθλητισμό επηρεάζεται όλο και περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα. Δυστυχώ αυτό είναι γεγονό και το είπατε, πρόκειται για εμπόριο νέων, ε, για ατασταλίες, ε, λαθροχειρίες, θα, βεβαίως οι ομοσπονδίες αθλητικές μόνες τους δεν έχουν τις αρμοδιότητες ε, να δράσουν ε, και να ασχοληθούν με το θέμα. Η πρωτοβουλία ευρωπαϊκή λοιπόν επιβάλλεται. Έχουμε ήδη μέσα νομοθετικά, έχουμε οδηγίες, ε, αρκεί να υπενθυμίσουμε μερικά σημεία που μας φαίνονται σημαντικά και που μας επιτρέψουν να δράσουμε. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα κριτήρια που ισχύουν για όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι η ιδέα μιας άδειας, μιας αδειοδότησης ε, είναι για αυτούς τους μάνατζερ. Μπορούν οι ομοσπονδίες να επιβάλλουν με τέτοια άδεια. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε, ένα σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε έναν συντονισμό παραδείγματο χάρη εκτός από τους ελέγχους και δεύτερο δυνατό μέτρο μια πλήρης διαφάνεια των ροών χρημάτων των, ε, που κυκλοφορούν σε αυτό το κύκλο σε αυτό το κύκλο κύκλωμα διότι είναι η πρώτη πηγή ε, διαφθοράς πρέπει να κάνουμε το παν για να αποφύγουμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που είναι σήμερα η πραγματικότητα. Και τρίτο σημείο που ανέφερε και η κυρία Πάκα, μια απαγόρευση δράσης για όσους αξιο... Ε, εκμεταλλεύονται τους ανήλικους, ανήλικες. Έχω... Έχουμε λοιπόν αρκετά μέσα, όπως είπατε και εσείς κυρία Επίτροπε, στη διάθεσή μας για να ζητήσουμε από τις Ομοσπονδίες ε, να κάνουν τώρα το παν για να δράσουν σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή το 2007 είχε ήδη λάβει υπόψη την έκκληση του Κοινοβουλίου για να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος από πλευράς αυτών των managers και εδώ στην μελέτη γίνονται πολύ καλές προτάσεις. Άκουσα ότι είστε διατεθειμένοι να περάστε στην παραπάνω ταχύτητα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις των managers των ποδοσφαιριστών μας είπαν ότι ζητούν ε, και οι ίδιες και οι ίδιοι να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε ό,τι είναι σάπιο να εξαλειφθεί όλα αυτά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον καλό ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χόνιμπολ θα λάβει τον λόγο για τη σοσιαλιστική ομάδα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε τυχεροί, υποθέτω, για να μπορούμε να μιλάμε για αυτή την πλευρά του παγκόσμιου πρωταθλήματος, διότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα καταδεικνύει περισσότερο από οτιδήποτε πόσο σημαντικό είναι το άθλημα αυτό, τα αθλήματα, το ποδόσφαιρο σε εκατομμύρια πολίτες, πόσοι παρακολουθούν με ιδιαίτερη χαρά και πάθος αυτό το άθλημα και λόγω αυτού είναι τόσο σημαντικό να διασφαλίσουμε ουσιαστικά ότι αυτό το άθλημα, το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα θα ρυθμίζονται όπως πρέπει <clears throat> και έτσι σε σχέση με τη δράση αυτή που έπρεπε να ληφθεί θα διασφαλιστεί σε σχέση με εκπροσώπους παικτών. Και δυστυχώς βλέπουμε κάποια πάρα πολύ σοβαρά θέματα και ολιστήματα, καταχρήσεις ε, πλήσιμου χρησίματος, ε, ε, εκμετάλλευση παικτών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά αδικήματα, εγκλήματα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση που μετά από τόσο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει τώρα. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή η συγκυρία από το ότι σήμερα όπου όλος ο κόσμος έχει επικεντρώσει την προσοχή του σε αυτό το άθλημα, στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια για τους ε, μεταρρυθμιστές ε, θα λάβει τον λόγο η κυρία Μακλάρεν παρακαλώ. Thank you, President. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως υποστηρίζω την πρωτοβουλία αυτή για να γίνει πιο διαφανή η δραστηριότητα των managers αυτών και θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυτό. Πρέπει ε, να ε, δούμε ότι τα θέματα όπως η διπλή εκπροσώπηση υπάρχει στην, στην ίδια ε, οργάνωση και όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Αλλά οποιαδήποτε νομοθεσία υπάρχει για τη ρύθμιση αυτής της δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τις εθνικές αθλητικές αρχές. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, επιβάλλει ρυθμίσεις στον κόσμο του αθλητισμού. Θα πρέπει να παρεμβαίνουμε μόνο εκεί όπου μπορούμε να οδηγήσουμε σε περισσότερη σαφήνεια. Σας ευχαριστούμε κυρία Μακράκιν. Ολοκληρώνουμε αυτό το γύρο με την παρέμβαση της κυρίας Βεζά. για ένα λεπτό εξ ονόματος Ενωτικής Αριστεράς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την ερώτηση που έθεσε η, η ε, πρόεδρος μας αυτήν την περίοδο ε, του παγκοσμίου κυπέλου. Καταγγέλλονται εδώ οι απειλές πάνω στην ηθική του αθλητισμού βασιζόμενοι σε ε, χιλιάδες εθελοντές που επιτρέπουν να ζήσει το αθλητικό πλεύμα έτσι όπως μας αρέσει διότι επιτρέπει την προσωπική άνθηση. Το κράτος όμως πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις όταν ε, πρόκειται για παρεκτροπές. Οι παρεκτροπές που είναι του ε, επαγγελματικού αθλητισμού, του business, εκεί όπου οι αθλητές ε, γίνονται εμπορεύματα και οι managers γίνονται μεσολαβητές, γίνονται μεσίτες που τοποθετούν αυτά τα προϊόντα, λαμβάνουν αστρονομικά ποσά ε, και οι ανήλικες ε, την χάνουν κακό μεταχείριτης. Ε, έχουμε τρελό χρήμα και οι, βεβαίως οι κυρώσεις είναι αυστηρές και τις ενίσχυσαν το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να βοηθήσουν. Ναι, κυρία Επίτροπε, πρέπει να δράσουμε και εγώ λυπούμαι που η Γαλλία ψήφισε μια αντίθετη νομοθεσία. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κυρία Βέζια. Ολοκληρώσαμε και αυτό το γύρο. Και τώρα ατομικά για 1,5 λεπτά ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όταν πριν αναφέρθηκε ότι ήταν λέει καθυστερημένη η ώρα να συζητάμε θέματα γυναικών μια και είχε φτάσει περίπου η ώρα μεσάνυχτα τώρα συζητάμε θέματα αθλητισμού αλλά τουλάχιστον συζητάμε αυτά τα θέματα δεν είχαμε ευκαιρία παλιότερα τώρα έχουμε και τώρα πρέπει αυτό να, το, να δραθούμε αυτή τη ευκαιρία. Είναι σημαντικό ότι τώρα κάνουμε λόγο για νέους νέους αθλητές και εκπροσώπους παικτών και τις δράσεις τους. Όπως αναφέρθηκε από πλευράς εισηγήσεως, υπάρχουν πολλά που αναμένουν εδώ είναι χρήματα που θέλουν να κερδίσουν σε σχέση με τη σταδιοδρομία τους, εγκαταλείπουν τα σχολεία, τις οικογένειές τους και μετά από κάποιο χρόνο περίπου ξαναβρίσκονται στο δρόμο. Και έχουμε εδώ και την πλειοψηφία αυτών των νέων που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα εμείς εδώ στην Ευρώπη έχουμε μια ευκαιρία κάτι να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε την ευκαιρία να επιβάλλουμε κυρώσει, να προστατέψουμε τους νέους εναντί τέτοιων καταχρήσεων και παραβάσεων. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα διάφορα αθλήματα στις διάφορες χώρες και να δούμε το συνολικό πρόβλημα. Τι πρέπει να γίνει προς όφελος αυτών των αθλητών και των αθλημάτων γενικά. Ευχαριστώ λεπτό. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ένα λεπτό η κυρία Μπόσκουρη Μποσκούρτ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Μποσκούρτ. Είναι μια, θα έλεγα, ασίδωτη δράση αυτή και δεν υφίσταται κανόνες. Και εδώ είναι ένα είδος εμπορίου ανθρώπων. Έχει εξεταστεί αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διαπιστωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει όμως κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ έχουμε και το θέμα του ευάλωτου χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων, των ανήλικων. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε χαρακτηριστικά ε, εμπορίου. Πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα έχει συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλλει. Πρόκειται για συγκεκριμένες διατάξεις για ε, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και καλύτερη ρύθμιση και διατάξεις από πλευρά των κρατών μελών και των λεσχών που, ομάδων, ποδοσφαιρικών ομάδων και συλλόγων που δεν ελέγχουν την κατάσταση σήμερα. Θα πρέπει η κατάσταση της άγριας δύσης, της ασυδοσίας και παρανομίας που υπάρχει να τερματιστεί. Πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχουν και δικαιώματα ανήλικων παικτών που πρέπει να διασφαλιστούν και πρέπει αυτοί να προστατεύονται πάντα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ συνάδελφε. Στον γύρο του Catch the Eye δύο συνάδελφοι έχουν εγγραφεί. Πρώτα ο κύριος Ματούλα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία του συναδέλφου Μπελέτ ε, για ένα νέο σύστημα που θα προστατεύει τα συμφέροντα των αθλητών ε, και θα ρυθμίζει τις δραστηριότητες των μάνατζερ ε, και θα εξασφαλίζει σωστή λειτουργικότητα στον τομέα αυτό τις μυστικές ε, προμήθειες ε, και λοιπά ε, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όχι μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και άλλα αθλήματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε σήμερα 6.000 μάνατζερ που αντιστοιχούν σε 30 διαφορετικά αθλήματα με ένα κύκλο εργασιών 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστημα θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί ένας ε, ε, ε κανονισμός, μια νέα ρύθμιση για όλους ε, και να ρυθμιστούν οι ευθύνε όλων αυτών. Μπόρις, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θετικό στοιχείο σε αυτή την ε, σε πολύ προχωρημένη ώρα συζήτηση αυτό το οποίο κάνουμε είναι η συνθήκη της Λισαβόνας που έχουμε στα χέρια μας και που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και μάλιστα υποχρέωση να παρέμβουμε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Σύντομα θα έχουμε και ε, την αντιμετώπιση αυτών των ε, αθλητικών ε, θεμάτων όσον αφορά την Πολωνία και γι' αυτό με ικανοποιεί αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις και διατάξεις. Το σύστημα δεν είναι διαφανές. Υπάρχει μεγάλη κατάχρηση και υπάρχουν πολλές παραβάσεις και παραβιάσεις. Και εδώ είναι πραγματικά δεινή η θέση των αθλητών, των παικτών. Έχουμε ε, συναλλαγές για τις μεταφορές, εξαγορές παικτών, τεράστια κονδύλια διακυβεύονται και βλέπουμε ότι υπάρχουν και υπερχρεωμένες ομάδες. Ε, Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Διακόπτεται. Η κυρία Επίτροπος Βασιλείου θα λάβει τον λόγο. Ας δούμε αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Αν γίνεται κάτω από τέσσερα λεπτά, τότε φτάνουμε μέσα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και όλοι συμφωνούμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι πολύ απολαυστικός για όλους μας. Σας ευχαριστώ όλους ε, πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας και τις προτάσεις σας που θα ληφθούν σοβαρότατα υπόψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποια δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, επιθυμητή. Οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν έχουν την εξουσία για να παρεύουν σε ορισμένες από τις χειρότερες περιπτώσεις κακής πρακτικής. Και τέτοιες πρακτικές αποκτούν ε, διεθνή ε, διάσταση καθώς γίνεται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένος ο αθλητισμός. Η επαγγελματικοποίηση και η διεθνοποίηση ε, του αθλητισμού ε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να δοθεί λύση σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο για να εξασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση στο θέμα των μάνατζερ. Παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τι νέε αρμοδιότητε που απέκτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Ε, πολλοί από αυτού που ασχολούνται με το αθλητικό κίνημα θα, θα δεχτούν ευνοϊκά μια τέτοια προσέγγιση προσέγγιση. Και θα πρέπει φυσικά να συνεργαστούμε στενά με τι ε, αντίστοιχε αθλητικέ ομοσπονδίε. Όπω ξέρετε, σκοπεύω πολύ σύντομα να, δημοσιεύσω, μια ανακοίνωση για τον αθλητισμό, η οποία σίγουρα θα αναφέρεται ε, με περισσότερε λεπτομέρειε στο θέμα αυτό. Θα ήταν λάθο να προδικάσω το αποτέλεσμα των ε, διαβουλεύσεων που θα πρέπει να κάνουμε και με εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώ επίση και με το αθλητικό κίνημα. Ε, θα περιμένω λοιπόν ε, να συνεργαστούμε